εδώ η συζήτηση. Ψηφοφορία αύριο 6 ώρα το απόγευμα. Θα ακολουθεί τώρα η έκθεση Ογιουλάντ ε, για περιορισμούς ε, θεώρησης ε, διαβατηρίων για Ρώσους αξιωματούχους που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση Σεργέη Μανίτση. Τον λόγο έχει η κυρία Όγιουλαντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το είναι πολύ γνωστό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το όνομα Σεκνέη Μακνισκή. Ήταν ο Σεπτέμβριο 2010 τότε που εγκρίναμε την ετήσια έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητήσαμε ε, δικαιοσύνη για αυτό τον θαραλέο Ρώσο ε, δικηγόρο που πέθανε πολεμώντα τη διαφθορά. Παρότι ο πρόεδρο Δημήτρη ε, ε, υποσχέθηκε ότι θα ρίξει φως αυτή την ε, υπόθεση δεν δόθηκε φως και την προηγούμενη εβδομάδα πολύ μικρή είναι η πρόοδος ανάμεσα σε έξι άτομα που εμπλέκονται για το θάνατό του έχουν απλώς κατηγορηθεί δύο γιατροί της φυλακής για αμέλεια Πέρασαν χρόνια από τον τραγικό θάνατο του Σεργέη Μπακνίσκη στη φυλακή μετά από ε, βασανιστήρια και χωρίς ιατρική περίθαλψη. Αυτό θυμίζει την περίπτωση του Βασίλη Αλεξανιά, ένα νέο ε, νεαρό δικηγόρο του Μιχαήλ Κοντροκόφσκι, ο οποίος πέθανε παράνομα στη φυλακή. Αντί να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν και κατέχουν τις θέσεις τους. Ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξοδεύουν τα βρώμικα λεφτά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγοράζουν έχουν ακίνητη περιουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μορφώνουν τα παιδιά τους. Εδώ ζητάμε το κράτη-μέλη να σταματήσουν την πρακτική αυτή. Αυτά πρέπει να αποτελέσει συγκεκριμένη αντίδραση σε αυτή τη συμπεριφορά και να δείξει την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζεται σε αξίες. Πρέπει να επανέλθουμε στις δημοκρατικές φιλελεύθερες αξίες μας και στην ένωμη τάξη. Σύμφωνα με την διεθνή διαφάνεια, η Ρωσία μαζί με την Ιγυρία βρίσκονται στον, στο τέλος του καταλόγου. Είναι λοιπόν εξαιρετικά υπεροπτικό εκ μέρους του Πούτιν να ζητά την, απελευθε... φιλελευθέρωση ε, των ε, κατόχων των νέων ε, διαβατηρίων που κατέχουν τα στελέχη της διοίκησης. Πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι οι αφέντες της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ δίπλα μας συζητήθηκε η κατάσταση στη Ρωσία. Αντί να σεβαστεί τους κανόνες της, ε, του, τη Συμβουλή της Ευρώπης οι Ρώσοι επέκριναν τη λεγόμενη ε, παρέμβαση στα εσωτερικά της Ρωσίας. Επίσης ε, απείλησαν ότι θα σταματήσουν να χρηματοδοτούν το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και όχι μόνο ε, εδώ, εδώ δεν είναι μόνο θέμα σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας αλλά είναι και το θέμα του διαλόγου γιατί η συμμετοχή της Ρωσίας στον ΠΟΕ δείχνει για μία ακόμα φορά ότι δεν έχουν σημασία για αυτούς οι κοινοί κανόνες παίρνει τον ΠΟΕ αλλά καρτ, κατά το δοκούν η Ρωσία. Αλλά είμαστε σαφείς. Η θέση του Μαγνίτσκι δεν είναι απλώς η τραγωδία ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει το οργανωμένο έγκλημα. Η προσωπική του μοίρα αντικατοπτρίζει το πόσο σύνθετη είναι η οργάνωση της ε, στην ρωσική κοινωνία. Η υποβάθμιση των θεσμών έχει οδηγήσει σε τεράστια διαφθορά και ε, επαναδραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Καθώς η Ρωσία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και η κοινωνία των πολιτών επιδιώκει το κράτος δικαίου, δεν μπορούμε να αφήνουμε τις τράπεζες Ευρωπαϊκής Ένωσης να δέχονται τις περιουσίες διεφθαρμένων ανθρώπων που κλέβουν από, την από τη Ρωσία. Από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το θέμα των ψηφισ... ψηφίσματα ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία θα πρέπει να, κάνουν, να τα κάνουμε πράξη και θα ήθελα να ζητήσω τους συναδέλφους αύριο να ψηφίσουν υπέρ αυτής της πρότασης. Σας ευχαριστώ κυρία Όγιουλαντ. Περνάμε στη διαδικασία Kids DI. Δίνω πρώτα απ' όλα το λόγο στον κύριο Μικολάσικ. Mm. Κύριε Μικολάσικ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν, είχα, δεν άκουα σωστά το όνομά μου και γι' αυτό δεν αντέδρασα αμέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Σεργέη Μαγνίτσκι είναι μαχητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν μαχητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το γεγονό ότι πολέμησε το οργανωμένο έγκλημα ε, δείχνει ότι έκανε έναν αγώνα για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό πρέπει να το στηρίξουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στηρίξει τη θέση αυτή και θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Ρωσία. Τέτοιου είδους συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες της είναι απαράδεκτη. Δεν είναι δημοκρατική χώρα αν δεν προσφέρει ιατρική βοήθεια σε ανθρώπους που τη χρειάζονται. Αν ένας φυλακισμένος ε, υπόκειται κακομεταχείριση και μετά τον αμελούν, στις ε, διαπραγματεύσεις με την Ρωσική Ομοσπονδία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπενθυμίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ κύριος Μεγκάλσικη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Μικολάσικ. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε, αλλά ο κύριος ε, Μαγνίσκη δεν αγωνιζόταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένας απλός άνθρωπος ήταν, ο οποίος ύψωσε το ανάστημά του. Ε, γι' αυτό παρενοχλήθηκε και πέθανε στη, σε ε, ρωσική φυλακή. Είναι λοιπόν το καθήκον μας να θυμίζουμε τη μοίρα όλων αυτών των απλών ανθρώπων στη Ρωσία που δεν θέλουν να ε, εμπλακούν σε αυτή τη διαφορά. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παγώσουν τα περισσιακά στοιχεία όσων ε, εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο θάνατο αυτού του ιδιαίτερου ανθρώπου ο οποίος ήθελε να είναι ηθικός ενώ στη χώρα αυτή βασιλεύει η ανηθικότητα. Αν είμαστε σοβαροί για τις ευρωπαϊκές αξίες, ε, για το πώς προχωράμε, θα πρέπει να φροντίσουμε τέτοια αδικία να μην επαναληφθεί. Σας ευχαριστώ. prywatnej... Θα ξεκινήσω με μια πολύ προσωπική σκέψη. Γεννήθηκα σε μια πόλη όπου ήταν εγκαταστημένοι Ρώσοι στρατιώτες. Γι' αυτό έχω συνειδηθεί με πολλούς κανονικούς Ρώσους. Είναι έντιμοι και καλοί άνθρωποι. Και ως Ευρωβουλευτής ε, είχα τη δυνατότητα να συναντηθώ με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης στη Ρωσία και ανθρώπους που δεν ήταν ίσως στην πρώτη γραμμή, αλλά οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία της αλλαγής στη Ρωσία. Σε μια πιο, για μια πιο δημοκρατική ευρωπαϊκή Ρωσία. Και πρέπει να πω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Μια χώρα που βρίσκεται στην Ευρώπη, που θέλει να την αντιμετωπίσουν ως ευρωπαϊκή, όπως αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιτρέπει τέτοιες πρακτικές. Πρώτον, την διεφθορά στο σύστημα δικαιοσύνης, αλλά και τέτοιες μεθόδους για την μεταξαφάνιση των ανθρώπων, όπως είπε ο κ. Μικαέλσκι. Ανθρώπων που θέλουν να είναι έντιμοι, ειλικρινείς δεν είναι μεγάλοι ηγέτες αντιπολίτευση, είναι απλή καθημερινή έντιμη άνθρωποι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρωτοσίβιτ. Τελείωσε η διαδικασία Catch the Eye και για να ολοκληρωθεί η συζήτηση θα ακούσουμε τον Επίτροπο, τον κύριο Πίμπαλξ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να λάβω μέρος σε αυτή τη συζήτηση για την περίπτωση Μαγνίτσκι εκπροσωπώντας την ύπατη εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο. Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για κοινούς περιορισμούς βίζας για τους Ρώσους Εξωματήχους της υπόθεσης Μαγνίτσκι είναι σημαντική πρωτοβουλία. Το Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια κινητοποιείται ειδικά από το ψήφισμα της 16 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι τις πάρα πολλές αγροάσεις που έχει οργανώσει και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες μαρτυρούν τη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη στην περίπτωση Μαγνίτσκι. Οι πρωτοβουλίες αυτές επίσης ε, προωθούν την κοινή μας προσπάθεια για να ασκήσουμε επίσης αρχές της Μόσχας για να διερευνήσουν την υπόθεση και νομοποιούν περαιτέρω την πίεση που πρέπει να ασκήσουμε στη Ρωσική Ομοσπονδία για να υπάρξει μια κατάληξη στην υπόθεση Μαγνίτσκι. Η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Κομισιόν ζητά επιμόνως από την Ρωσία να υπάρξει μια σωστή έρευνα και βεβαίως θίγουμε αυτό το θέμα σε όλες τις επαφές μας με τις ρωσικές αρχές. Μάλιστα, η περίπτωση Μαγνίτσκι είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη των εξαμηνιαίων συναντήσεων μας και επίσης θίγεται τακτικά σε επίπεδο υπουργών και στη Σύνοδο Κορυφής. Τον περασμένο μήνα η Βαρόνη Άστον αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην περίπτωση Μαγνίτσκι όσον αφορά μάλιστα την πολιτική χρήση της δικαιοσύνης και σημείωσε την ανησυχία που υπάρχει για το ότι δεν υπάρχει πρόοδος στην υπόθεση Μαγνίτσκι, κάτι το οποίο αποτελεί μέρος των γενικότερων εξελίξεων στη Ρωσική Ομοσπονδία, κάτι το οποίο ανισχύει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση η ομιλία και η συζήτηση που ακολούθησαν αναφέρθηκαν στον ρωσικό τύπο. Τον Απρίλιο φέτος ο πρόεδρος Φαν Ρόμπαϊ ε, έγραψε μια επιστολή στον ε, πρόεδρο Μετβέντεφ ειδικά για την υπόθεση Μαγνίτσκι και ανέφερε τρία σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, ζήτησε από τη ρωσική κυβέρνηση να υπάρξει μια κατάληξη σε αυτή την υπόθεση. Δεύτερον, ζήτησε από την Ρωσία να σταματήσει με τα θάνατον δίωξη του κυρίου Μαγνίτσκι και τρίτον, ζήτησε να τερματιστεί ο εκφοβισμός της μητέρας και της χήρας του κυρίου Μαγνίτσκι. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης συνεχίζει να υπενθυμίζει αυτό το ζήτημα, αλλά δεν έχουμε λάβει απάντηση στην επιστολή. Όλα αυτά, καθώς και η απάντηση η οποία δεν έχει δοθεί στην επιστολή του Πρόεδρου Φαν Ρόμπαϊ, επαναλήφθησαν τελευταία από την Επίτροπο Μάλμστρομ στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Εσωτερικών που έλαβε χώρα στις 22 ε, Σεπτεμβρίου στη Λευκοσία παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα και θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε για τρεις πολύ καλού λόγους. Πρώτον λόγω της φύσης της υπόθεσης. Είναι μια περίπτωση ενός Ρώσου πολίτη, δικηγόρου, νεαρού πατέρα, ο οποίος συνελήφθη και κακοποιήθηκε από αστυνομικούς γιατί αντιστάθηκε στην απάτη και την κατάχρηση εξουσίας ε, από αξιωματούχους. Πρόκειται λοιπόν για βαριά παραβίαση του νόμου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις βασικές αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του κράτους δικαίου, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα τα υπερασπιστούμε αυτά. Η περίπτωση Μαγνίτσκι έχει γίνει μια εμβληματική περίπτωση και υπόθεση όχι μόνο για τους Ρώσους αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση Μαγνίτσκι είναι επειδή θεωρούμε πως και η ίδια η Ρωσία θα πρέπει να επιλύσει αυτή την υπόθεση γιατί συμβολίζει την κατάσταση της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Οι επιχειρηματίες το θεωρούν την Λιδία λίθο για την σταθερότητα και την πρόβλεψιμότητα της Ρωσίας ως επενδυτικό προορισμό καθώς δεν είναι μια πολύπλευρη ε, περίπτωση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφθοράς. Καταβάλλονται προσπάθειες λοιπόν κατά της διαφθοράς όσον αφορά τον εξυγχρονισμό της Ρωσίας και βεβαίως το να λυθεί αυτή η υπόθεση θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε εταίρους και επενδυτές πως η Ρωσία παίρνει στα σοβαρά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τρίτον, είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει στα σύνορά της μια σταθερή, ε, δημοκρατική και οικονομικά βιώσιμη Ρωσία με ένα κράτος δικαίου. Αυτά τα οποία είναι σημαντικά για να ενταχθεί η Ρωσία σε ένα παγκόσμιο σύστημα με κανόνες όπως παραδείγματο χάρη η ένταξή της στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Περιπτώσεις όπως αυτές, ε, όπως η υπόθεση Μαγνίτσκι δυστυχώς δεν βοηθούν σε αυτό το κλίμα. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν είναι συγκεκριμένη δράση από την πλευρά της ρωσικής κυβέρνησης, μια σαφής απόφαση για να ερευνηθεί σωστά η υπόθεση Μαγνίτσκι και να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Οπότε σημειώνουμε την σύστασή σας που απευθύνεται προς το Συμβούλιο για περιοριστικά μέτρα σε Ρώσους αξιωματούχους που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση. Μαγνίτσκι στέλνει ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα. Βεβαίω το να δράσουμε, να κάνουμε κάτι απαιτεί ομοφωνία από όλα τα κράτη-μέλη. Και πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία όσον αφορά τη σχέση μας με την Ρωσία. Περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ ευαίσθητο και λεπτό μέσο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης. Επιπλέον τα περιοριστικά μέτρα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέρος μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα περιλαμβάνει και πολιτικό διάλογο και συμπληρωματικές προσπάθειες. Σας διαβεβαιώ πως η υπόθεση Μαγνίτσκι θα παραμείνει ψηλά στις ε, επαφές μας με την Ρωσία. Οι δε κυρώσεις πρέπει να παραμένουν το τελευταίο μέσο που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλιώς θα γίνουν το μόνο μέσο στις σχέσεις μας όταν διαπράττονται τέτοια εγκλήματα. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, να επαναλάβω ακόμη μία φορά εκ μέρους της ε, Βαρόνης Άστον πώς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση Μαγνίτσκι και να θέτουμε το ζήτημα στις ρωσικές αρχές σε κάθε ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Τελείωσε εδώ πέρα η συζήτηση. ψηφοφορία αύριο 6 ε, ώρα το απόγευμα. Επόμενο σημείο, έκθεση Μορέιρα για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ο εισηγητής έχει το λόγο για 4 λεπτά. Ε,